Okay. Good morning. Καλημέρα σας. Ich darf die Καλημέρα συνάδελφοι. Ξεκινάει η συνεδρίαση της 27 Μαρτίου. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι είναι δημόσια η μετάδοση και στο διαδίκτυο της συνεδρίασής μας. Ξεκινάμε πάλι σήμερα με τις ψηφοφορίες και θα ήθελα καταρχά να σας ενημερώσω ότι και σήμερα ότι σήμερα μάλλον ε, θα μας ε, συνοδεύσει ένας δημοσιογράφος ο οποίος γράφει ένα άρθρο για το έργο μου ως ε, Πρόεδρος της Επιτροπής, ε, χαιρόμαστε πάντα όταν το έργο της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των, ε, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταδίδεται και δημοσιεύεται. Και τώρα να περάσουμε σε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά αν θέλετε να ψηφίσουμε. Να ελέγξουμε κατά πόσο λειτουργεί το σύστημα. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. 20 ψήφοι, αν και είναι 23 ε, οι παριστάμενοι. Παρ' όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε. Ja. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Να περάσουμε στο 8. Προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολέμηση τη απάτη, αντίτηση έκθεση 2010. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 3 το ψηφίζουμε, το 2 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 5. Με προφορική τροπολογία. 5 έως 10. Να ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ, γιατί 5 έως 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Να επαναλάβουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλιστα να ήταν σαφέ τώρα. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 21 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Σαφές, το αποτέλεσμα εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 με σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 Α, θέλετε να το αλλάξουμε. Α. Α, συνολικά μέχρι την 25, ε, αν συμφωνείτε. 26 έως 25, μαζί. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Τροπολογία 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31. 31 έως 29 από κοινού, αν συμφωνείτε, μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ, γιατί 34. Έναρξη ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Από. Αποχές. Δεν είναι σαφές και αυτό να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε μου φαίνεται οριακό το αποτέλεσμα. 37 παρακαλώ, να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Έναρξη ψηφοφορία, αν ψήφισατε όλοι, πέρα. Α, ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 στα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Οριακό το αποτέλεσμα, παρακαλώ ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 41. 41 έως 45 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Είκοσι ψήφοι υπέρ, μία αποχή εγκρίνεται. Και περνάμε στο 9 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Απαλλαγή 2010 Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο. Έχεις. Okay, ich hatte gerade von unterrichtet, dass zwei Änderungsanträge zurückgezogen Έχουν αποσυρθεί δύο τροπολογίες με ενημερώνουν, η 6 και η 36. Η 6 και η 36 έχουν αποσυρθεί. Dann können wir... Άρα, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Οι 5, 2, 3, 4 και 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η 6 αποσύρθηκε, η 7 λοιπόν υπέρ. Κατά, αποχές, να το ελέγξουμε αν θέλετε γιατί είναι 7. Έναξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα να ψηφίσουμε την απόφαση ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, και περνάμε έτσι στην 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 12 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε αν θέλετε για την 12 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πέρας Ήταν ωριακό το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Η 12. Η 13 τώρα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελεκτρονικά για το 14 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 18 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι σαφές. Δεν παρακαλώ. Και τώρα πάμε στην επόμενη υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Για την 17 υπέρ, ε, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται, αλλά δεν ε, σηκώσατε όλοι τα χέρια σας. Εγκρίνεται άραγε. Πέρας. Ναι, σας παρακαλώ να συμμετέχετε στην πρωινή γυμναστική. Γιατί έτσι είναι οι ψηφοφορίες, τι να κάνουμε. Και τώρα περνάμε στην 17, λέει ο πρόεδρος. Α, όχι, την ψηφίσαμε την 17. Ναι, λες και να θέλω να την ψηφίσω. 20, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 σε τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. 27 και 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινονται. Η 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 29 καταπίπτει. Η 31 έως 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται αλλά στο ελέγξουμε για σιγουριά. Ηλεκτρονικός έλεγχος η 31 έως 34 πέρας ψηφοφορίας όχι, ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Η 36 αποσύρθηκε, η 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 37 υπέρ, να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 35 παρακαλώ. Έναρξη ψηφορία για την 35. Πέρας. Απορρίπτεται. Αυτό δεν είχα πει, ότι απορρίπτεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, 2 κατά εγκρίνεται. Πολύ σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο Γενικό Προϋπολογισμό του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματο. απόφαση, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, αποφασίζεται, συνολική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. παράγραφος 12, τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. <coughs> τροπολογία 4, σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του ψηφίσματος αποτροποποιήθηκε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας υπέρ. Μάλλον έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, σαφέστατα. τώρα αλεκτικό συνέδριο. Στο 11 της ημερήσιας διάταξης. Τροπολογία 1 και 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο της απόφασης ε, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 5. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ή 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α, συγγνώμη, υπορρίπτεται να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε για τη 10 παρακαλώ για τη 10 ελέγχουμε ηλεκτρονικά τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 15 σε δύο τμήματα υπέρ. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπέρ. δύο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 16 και 17 θέλετε να τις ψηφίσουμε μαζί. Α, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Οι 16 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Πάμε τώρα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Όχι. Α, ναι. Λέει ο Πρόεδρος. <laughs> Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τροπολογία 4, 2 και 3. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε παρακαλώ έναξη ψηφοφορία. αν ψηφίσατε όλοι πέραση ψηφοφορία απορρίπτεται τροπολογία 5 και 6 Αν απορριφθούν οι άλλες εγκρίνονται. Χθες το εγκρίναμε επειδή απορρίψαμε τις άλλες. Ήθελα και χθες να σας ρωτήσω. Όταν λέτε ότι κατά συνέπεια εγκρίνονται, ποιος το αποφασίζει αυτό η γραμματεία? ξέρω, θέλετε να ψηφίσουμε, οπωσδήποτε. Ήθελα α, απλά να ξέρω από πού μπορεί να μας κυνηγήσουν, καταλαβαίνετε. Ναι, είναι πάντα δύσκολα όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, λέει ο Πρόεδρος. ναι, ναι, ναι, μου κάνει πλάκα η κυρία Γκρέσλε και με ρωτάει αν είναι το δίκαιο της ε, Κομόπολης από την οποία προέρχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, συνάδελφο Ινια Γκρέσλα και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να το ελέγξουμε παρακαλώ δεν την 8. Ψηφίσατε όλοι. Αν δεν ψηφίσατε... Α, ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 9 σε δύο τμήματα υπέρ το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 14 και 15 καταπίπτουν, οι 16 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 16. Αν ψηφίσατε όλοι, να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Ναι, 13 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται και καταπίπτουν λοιπόν οι 17, 18 και 19. Συνεχίζουμε με την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 22, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. Ναι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 23, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θεωρώ ότι εγκρίνεται. 24, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα η 30 και η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 32 έως 35 και συνεχίζουμε με 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ, Παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 36 και την 37 μαζί. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 38 και 38 λοιπόν καταπίπτουν 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 41 σε δύο τμήματα παρακαλώ το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σύνολο ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 44. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 44 παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Ίσως να έκανε λάθος Ευτυχώ που προσέχει και η Επιτροπή. Το σύνολο της ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, εγκρίνεται. Επόμενο. Επιτροπή των Περιφερειών. Τροπολογία 5 και η 4. Υπέρ μαζί. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 3 και η 2 έχουν αποφασιστεί. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνολική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη. Τέλος. Σαφές και το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά. Η 6 τώρα, υπέρ. κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε για την 10 αν θέλετε ηλεκτρονικά πέρας σαφές το αποτέλεσμα εγκρίνεται Μα χαίρετε και ο συνάδελφος Στάς. Εγκρίνεται λοιπόν η 10 και περνάμε στην 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 14 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Πρώτο τμήμα, ε, δεύτερο τμήμα, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και η 15 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19, υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. ist geschlossen. Εγκρίνεται. Σαφέστατα. Και έτσι περνάμε λοιπόν στο 14. Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ολική ψηφοφορία τώρα, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορία. Αν ψηφίσετε όλοι. Τέλος. Πέρασε. Πρόλαβε και ο συνάδελφος. Για να επηρεάσει κρίσιμα το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο, το 15. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Τροπολογίες 1 και 2. Μαζί, ε? με την ε, γλωσσική τροπολογία της ισπανικής ε, μετάφρασης. Συμφωνείτε παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφ, ε, τώρα ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε την απόφαση παρακαλώ. Αν ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν η απόφαση. Τροπολογία 2 τώρα. Υπέρ. Από την Επιτροπή Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 1 και, την, και αυτή της Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4 λίμπε υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το σύνολο του ψηφίσματος και πάλι ηλεκτρονικά. Έναρξη πληροφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. So, Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την ε, γρήγορη ψηφοφορία. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές και για τη χθεσινή ημέρα γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να τους χειροκροτήσουμε και τα λέμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα πάλι. Σας ευχαριστώ. See you in the afternoon. Ich unterbreche die Sitzung. Eh? Yes, yes, yes, please. Uh, it's another room. Yeah. Uh, uh, ein äh, kleiner Hinweis. Μία μικρή υπόδειξη σήμερα το απόγευμα. Θα συναντηθούμε, θα γίνει συνεδρίαση σε άλλη αίθουσα. Παρακαλώ να το ελέγξετε. 5 5B00. In this building. Okay, it's PHS 5B01. Στον πέμπτο όροφο, σε αυτό το κτίριο. Don't forget your cards. Τις κάρτες μην ξεχάσετε. Thank you.